και όπως γνωρίζετε θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30 την έκθεση αυτή και τις τροπολογίες της. Θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Καταρχήν να σας πω ότι λάβαμε από το Συμβούλιο δύο θέσεις για πρώτη ανάγνωση που θα πρέπει να εγκρίνουμε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. Οι τίτλοι θα παρουσιαστούν στην παρούσα Ολομέλεια, στην παρούσα σύνοδο. Και η διαδικασία ξεκινάει από τις 26 Οκτωβρίου. Από τους πράσινους έλαβα ένα αίτημα διορισμού που ε, εντάσσεται στην παρούσα σύνοδο και εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται ο εν λόγω διορισμός ή διορισμοί. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση Γκάρτια Θάμπαλ Γκάρδια θαμπαλ ρουμπιαλ για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μέσα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδιαθάμπαλ, ο εισηγητής. Η κυρία μάλλον. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος. για τρίτη φορά παρεμβαίνω στην Ολομέλεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και τους γνωμοδότες Υπάρχουν τρεις ε, λόγοι για τους οποίους τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν απαραίτητο μηχανισμό για να φτάσουμε σε μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη διότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 οι δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί δραστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αντιμετωπίσαμε παράλληλα και την χρηματοοικονομική κρίση στα μέσα του 2008. Επίσης, η αγορά είναι πιο περιορισμένη και δεν υπάρχει πρόσβαση σε πιστώσεις και κεφάλαια ή στις κεφαλαιαγορές. Επίσης, η στρατηγική 2020 θα χρειαστεί 1,6 δις για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Γι' αυτό θα βοηθήσουμε τις επενδύσεις σε προγράμματα που θεωρούμε στρατηγικής σημασίας και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτές τις επενδύσεις εκεί που δεν προωθήθηκαν μέχρι τούδε. Έτσι θα βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία και θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πείρα μας από το 2000 και μετά και τις αξιολογήσεις που έχουμε μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας ε, του μέλλοντος. Μπορούμε να περιορίσουμε τα μέσα και τους μηχανισμούς, θα ε, διευρύνουμε την κρίσιμη ε, μάζα και θα διαφοροποιήσουμε τους κινδύνους σύμφωνα με μία προσέγγιση βάση χαρτοφυλακίου. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι πιο λογικό, το οποίο να μην επιβαρύνει διοικητικά τους ενδιάμεσους και να βοηθήσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές. Ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο θέμα είναι η ευελιξία αυτών των μηχανισμών που θα πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές τάχιστα. Γι' αυτό θα θέλαμε η δημοσιονομική αρχή, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να μπορούν να αλλάξουν το ποσό που προσδίδεται σε κάθε πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορούμε να πούμε ότι και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούμε ως προς τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων και ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Αυτή όμως η πρόταση ε, δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες, όχι μακροπρόθεσμες. Θα πρέπει να έχουμε ασφαλή και βιώσιμα μέσα έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα μέσω και μακροπρόθεσμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να βοηθήσουμε ε, την πορεία αυτή μέσω των επενδύσεων που πραγματικά πρέπει να πραγματοποιηθούν και να λάβουμε υπόψη τις ε, επενδύσεις που θα πρέπει να προωθηθούν μακροπρόθεσμα μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας 3 και Φερεγγιότητα 2. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει κάτι να μας πει σε σχέση με το πλαίσιο της Βασιλείας 3. Πιστεύω πως ναι. Επίσης και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα συμβαδίσουμε γιατί κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Επίτροπο και συνάδελφο και φίλο μπορώ να πω, τον κύριο Λεβαντόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά που σας απευθύνομαι σήμερα, δεν υπάρχουν υπουργοί σήμερα. Βεβαίως ε, στην Κομισιόν. Καλωσορίζουμε την έκθεσή σας, ε, κυρία Γαρδία Σάβαλ. Και βεβαίως ε, εδώ πέρα φαίνεται και η ικανότητά σας καθώς εξασφαλίσατε μεγάλη στήριξη ε, της έκθεσης σας και βεβαίως χρειαζόμαστε τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για έναν ενισχυμένο ρόλο για χρηματοδοτικά μέσα στις επόμενες δημοσιονομικές προεπτικές για ένα απλούστατο λόγο γιατί είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι και πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως το δυνατόν περισσότερο το κάθε ευρώ του προπολογισμού μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ακριβώς αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Και έχετε δίκιο, δεν αναπληρώνει αυτό τον προπολογισμό. Είναι ένας πολλαπλασιαστής αλλά δεν είναι στρατηγική μείωση ε, του προπολογισμού ούτε να αντικαταστήσουμε τις επιχορηγήσεις με δάνεια. Βεβαίω και τα δύο χρειάζονται και αυτό είναι το μήνυμά μας προς το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε κάποιους πολλαπλασιαστές ε, και να υπάρχει μια σχέση μεταξύ των αναγκών βεβαίως και των δυνατοτήτων, αλλά αυτό δεν αντικαθιστά τον προϋπολογισμό και ε, δεν είναι δυνατόν με δάνεια να αντικατασταθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Γιατί λοιπόν το χρειαζόμαστε αυτό γιατί το κενό νομίζω είναι εμφανές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια αποστροφή ε, του κινδύνου λόγω της ε, κρίσης και βεβαίως ε, σε αντίθεση με την άλλη όχθη του Ατλαντικού εδώ πέρα στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον ε, τραπεζικό τομέα και όχι από τις ε, αγορές. Γι' αυτό χρειάζεται να μειωθεί αυτή η αποστροφή του κινδύνου και να χρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα έργα, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, ε, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Και όσον αφορά τώρα τα ομόλογα έργων για τα πιλωτικά μας έργα, μπορώ να σας ανακοινώσω πώς υπογράφει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ακριβώς τέτοια έργα στις τρέχουσες μεσονομικές προοπτικές 2007-2013 και πάλι συμμορφόμενοι πλήρως με την ε, δήλωση πως θα πρέπει να καλυπτόμαστε από πάρα πολύ αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η Δημοσιονομική Αρχή πριν δώσει την έγκριση για την χρήση ενός χρηματοδοτικού μέσου θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερη και να υπάρξει και μια εξάντε αξιολόγηση αλλά και πλήρης παρακολούθηση των έργων και μια τελική έκθεση. Αυτό χρειαζόμαστε. Και ευελιξία. Επίσης κάτι το οποίο αναφέρατε στην έκθεσή σας. Χρειάζεται ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις διακυμάνσεις των αγορών και στο τοπικό περιβάλλον στις χώρες της Ένωσης. Αυτή λοιπόν είναι μια ανάγκη. Ο ενισχυμένος ρόλος των χρηματοδοτικών μέσων που χρειάζεται οπωσδήποτε για να γεμίσει το κενό μεταξύ των όσων χρειαζόμαστε για την Ευρώπη και των περιορισμένων πόρων που έχουμε στον προπολογισμό μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεισφορά σας και έτσι νομίζω θα βγούμε και θα οδηγηθούμε σε μια ανάκαμψη όταν αντικαταστήσουμε την λιτότητα με πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε ο Ζάμπιερ Οντί, εξ ονόματος της Επιτροπής Προπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη κυρία Ιβάνοβα η οποία είχε άλλε κοινοβουλευτικέ δραστηριότητε και η οποία μας, μου ζήτησε να σα ε, κάνω μια περίληψη της, ε, την έκθεση τη επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών. Έχει λάβει υπόψη του τη δυνατότητα μόχλευση και τι πολλαπλασιαστικέ επιπτώσει των νέων αυτών καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων αλλά έχουμε λάβει υπόψη μας την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και την ενίσχυση ενίσχυση του προσωπικού της Ένωσης για να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Το δεύτερο αφορά τις ε, χρηματοοικονομικές αγορές. Θεωρούμε ότι αυτά τα μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή μάλλον να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν δεν ε, υπάρχει αντιστοιχία όταν δεν υπάρχει ε, προσφορά από την ιδιωτική αγορά και λυπόμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη το θέμα των δια των δικτύων μεταφορών της Ευρώπης, τα οποία είναι επενδύσεις άμεσα αποδοτικές. Έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Αντώνιο Καντσάν, ο οποίος θα μιλήσει από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι δεν, μπολώ, δεν μιλώ με ακρονίμια, διότι πολλοί πολίτες μας παρακολουθούν και έχει μεγάλη σημασία να καταναούν περί τίνος πρόκειται, γιατί πράγμα μιλάμε. Γι' αυτό αναφέρομαι σε... και στις επιτροπές με τον πλήρη τους τίτλο. Έχει το λόγο ο κύριος Καντσάν, τώρα εξ ονόματος Επιτροπής Βιομηχανίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σκεπτικό ότι τα δημοσιονομικά μέσα είναι ανεπαρκή. Γι' αυτό οι λίγοι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας ε, δεν μπορούν παρά να αξιοποιηθούν μέσα στα πλαίσια των καινοτόμων μηχανισμών που είναι ειδικά ταμεία ή ε, ομολογίες έργου. Θα πρέπει λοιπόν να ενταχθούν στη συνδρομή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές και τα ενδυνάμει βιώσιμα σχέδια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κινηθούμε και πέραν από αυτό το πλαίσιο και να κινηθούμε με ομόλογα τα οποία ε, στην ουσία θα είναι δανειοδοτήσεις, μακροχρόνιες δανειοδοτήσεις. Εκεί έγκυται η πραγματική ανάπτυξη, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Το λόγο έχει η κυρία Κλέβα για δύο λεπτά για να γνωμοδοτήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι μια στήριξη υπομορφής, υπομορφή εγγυήσεων ε, δανείων ε, και λοιπόν μέσων. Μια λοιπόν ε, διάφανη εξέταση αυτών των ε, μέσων σημαίνει πως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εδώ πέρα την εισηγήτρια την κυρία Γκαρτία Σάβαλ γιατί έκανε δεκτές τις περισσότερες ε, τροπολογίες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και αφορούν την χρήση αυτών των μέσων στην πολιτική συνοχή. Μπορεί να παίξουν εκεί πέρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής ε, συνοχής. Μπορεί να υπάρξει έτσι μια αποτελεσματικότερη χρήση τους και να υπάρξει μια γρηγορότερη χρήση αυτών των μέσων. Νομίζω πως θα πρέπει να στηρίξουμε την Κομισιόν για μια πιο αποτελεσματική εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα στην επόμενη προγραμματική περίοδο, κάτι το οποίο μπορεί να ωφελήσει τις ε, επενδύσεις. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό τα μέσα αυτά να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς και στόχους ε, της ε, πολιτικής συνοχής, αρκεί βεβαίω να διασφαλιστεί παντού η διαφάνεια. Χρειάζεται λοιπόν ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει καθοριστεί πριν από την αρχή της νέας προγραμματικής περίοδου. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουν επιτυχία αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει να βελτιωθούν και οι τεχνικές δυνατότητες και στο επίπεδο της διοίκησης, αλλά και όσον αφορά τις τράπεζες και τους τελικούς χρήστες. Επίσης είναι σημαντικό αν είναι να αυξηθεί η χρήση τους, να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για όλους τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο του προπολογισμού της Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Κατά την παρέμβαση αυτή, κυρία Κλέβα, μου είπαν, μου κοινοποίησαν οι διερμηνείς ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Σας παρακολουθήσουν ο ρυθμός σας ήταν τόσο γρήγορος που ήταν αδύνατο να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λαμβάνετε υπόψη αυτό τον παράγοντα, διότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν οι διερμηνείς. Έληξε ο γύρος των παρεμβάσεων εξ των ε, Επιτροπών και τώρα έχουμε τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ έχει το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρτία Δαμπάλ για την εξαιρετική της εργασία και συνεργασία μαζί μας. Πιστεύουμε ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως μας πρότεινε η Κομισιόν, θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης για να υπηρετήσουμε την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη καθώς και την εξυγίανση των δημοσίων ε, οικονομικών, όπως ε, τόνισε και ο Επίτροπος. Πρόκειται για έναν μοχλό για την οικονομική μας ανάπτυξη τα βιώσιμα σχέδια δεν ε, λαμβάνουν πάντα χρηματοδότηση, γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε στα σχέδια τα οποία προσδίδουν μεγάλα ε, έσοδα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πολυσχεδία αυτά μέσα και παράλληλα να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό, το οποίο δεν γνωρίζει πάντα περί τίνος ε, πρόκειται. Δεν πρέπει να χαθούμε στο λαβύρινθο αυτής της οικοδόμησης. Θα πρέπει να, επίσης να υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος για την ε, χρήση και την ευελιξία αυτών των μέσων για να μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματική οικονομία για να είναι δελεαστικά για επενδύσεις. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο αυτών των μηχανισμών για την ανάπτυξη της κεφαλαίου στην Ευρώπη, αλλά δεν θα πρέπει να ε, διασυνδεθούν με περίπλοκα προϊόντα. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ, εξ ονόματος των σοσιαλιστών για δύο λεπτά και πάλι έχει το λόγο ο κύριος Γκέραν Φέρμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, την κυρία Κάρδια Θαβάλ, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά για, επί ενός πολύ σημαντικού θέματος για το μέλλον και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης δεν πρέπει να, να ασχολείται μόνο με τα κατεπήγοντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Όχι, πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προκτική για την οικονομία μας με επενδύσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη. Η κρίση δεν σημαίνει μόνο κατάρρευση των θεσμικών οργάνων και των τραπεζών. Ξέρουμε ότι συνεπάγεται και ένα πρόβλημα επενδύσεων. Για πολλά χρόνια έχουμε χαμηλό επίπεδο επίπεδο επενδύσεων και τώρα φτάσαμε σε τόσο χαμηλό σημείο που πλέον είναι επικίνδυνο. Ε, όπως επεσήμανε βεβαίως και η εισηγήτρια, οι επενδύσεις είναι τεράστιες και Χρήμερα υπάρχουν δυστυχώς μεγάλοι περιορισμοί στον κοινοτικό προπολογισμό, στου εθνικούς προπολογισμού. Οι τράπεζες έχουν πολύ αυστηρότερε τεχνικές προδιαγραφές και είναι δύσκολο να βρούμε χρήματα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε με καινοτόμο τρόπο διαφορετικά. Και παραδείγματο χάρη τα ομόλογα έργου είναι καλά παραδείγματα τα οποία θα δοκιμαστούν φέτο. Όπως ε, ανέφερα και εγώ στην προηγούμενη έκθεσή μου, νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει οι επιχειρήσεις να μπορούν να εκδώσουν εμπόλογα έργου ασφαλή και ελκυστικά. Τα, τα συνταξιωτικά ταμεία αντί να αφήνουν τα χρήματά τους να κοιμούνται σε κάποιο λογαριασμό, να τα χρησιμοποιήσουν επενδύοντας σε έργα υποδομής. Χαίρομαι πολύ που ο Επίτροπος είπε ότι αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, ότι μιλάμε για χειροπιαστά έργα τα οποία προετοιμάζονται, πρόκειται να υπογράψετε συμφωνίες φυσικά. Το Κοινοβούλιο θα αξιολογεί, θα παρακολουθεί και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερα ποσά και ενδεχομένως θα δοκιμάσουμε και κάποια άλλα μοντέλα που έχουν περισσότερες δυνατότητες. Πιστεύω ότι αν θέλουμε η Ευρώπη να φύγει από ε, την περίοδο της λιτότητας των περιορισμών, να μπει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, να, χρησιμοποιήσουμε τέτοια ε, έργα. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο η κυρία Γένσεν. E Κύριε Πρόεδρε, εδώ και πολύ καιρό είχαμε τονίσει το γεγονός ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική μέσω δανειοδοτήσεων και εγγυήσεων. Μας απασχόλησε επιμακρών αυτό το θέμα, γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η ανακοίνωση από πλευράς της Επιτροπής. Πολλά και άκρος ενδιαφέροντα προβάλλονται και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στα πλαίσια της ΕΤΕ υπάρχει, μάλλον ε, διαπιστώνουμε μια μεγάλη επιτυχία, πολλές επιτυχίες και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Χρειάζεται δημιουργία μεγαλύτερου κεφαλαίου για να φέρουμε σε πέρα σε διάφορα προγράμματα στον τομέα της, των ερευνών, υποδομών, καινοτομίας, μεταφορών. Πρόκειται για δύσβατα θέματα όπου έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τους κατάλληλους πόρους μέσω της ε, κεφαλαία αγοράς. Αυτό ελέγχθη από πολλούς ομιλητές και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να τονίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ανάπτυξη και απασχόληση. Περί αυτού πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα ευρύ φάσμα μέσων και έχει απόλυτο δίκιο η Επιτροπή επ' αυτού. Πρόκειται για καινοτόμα μέσα, τα οποία όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την παραδοσιακή μας πολιτική. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τους παραδοσιακούς μας προϋπολογισμούς και αυτό το τόνισε και ο Επίτροπος. Ως προς τη, τα ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων υπάρχει ένα πιλωτικό σχέδιο και ευρωπαϊκές εγγυήσεις έτσι ώστε στο τομέα μεταφορών και ενέργειας να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σχέδια εκδίδοντας ομολογίες. Μία παράλληλη αγορά υπάρχει και στις ΗΠΑ, γιατί συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα και ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να εγγυηθούν ρευστότητα με υψηλή απόδοση. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να προβούμε σε δοκιμές και να δούμε κατά πόσο αυτή η αγορά θα μπορούσε να προωθηθεί και μετά από λίγα χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε μια παρόμοια αγορά με αυτή που υπάρχει στις ΗΠΑ και έτσι να μην έχουμε άδεια ταμεία πλέον. Να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα διάφορα προγράμματα. Δεν, είναι δεν παρουσιάζουν όμως όλα το ίδιο ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και από τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για μία περιορισμένη επένδυση και δεν υπάρχουν κίνδυνοι έτσι ώστε να διονγκωθεί ο προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γένσεν εξ εκτός ε, των συντηρητικών. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Πορέμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων θα βοηθήσει την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ταλαιπωρείται από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τα, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της, καλής, της χρηστής διακυβέρνησης και να χρησιμοποιούν και μέσα όπως οι επιδοτήσεις. Θα πρέπει να διευκολύνουν την ε, υλοποίηση των έργων, να έχουν την απαραίτητη οριμότητα και να προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια σε έργα δημόσια υποδομή, ώστε να εγγυώνται την βέλτιστη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων. Το σημαντικό θα είναι εδώ ότι θα υπάρχει ένα απλουστευμένο νομικό πλαίσιο που δεν συνεπάγεται ένα επιπλέον βάρος για του ενδιάμεσου και του δικαιούχου, αλλά θα είναι ελκυστικό και για το δημόσιο και για του ε, ε, ιδιώτες επενδυτές. Ο φόβος είναι ότι αυτά τα, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν μόνο βραχυπρόθεσμα για ταχεία και κερδοφορία και ότι δεν θα συνεισφέρουν στην ε, και μακρο, στα βιώσιμα και μακροχρόνια έργα. Λίγη αυτός ο γύρος με την παρέμβαση για ένα λεπτό του κυρίου Μέρφυ εξ ονόματος της Γκουε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το υπόβαθρο εδώ πέρα της έκθεσης αυτής είναι η κατάρρευση των επενδύσεων σε ολόκληρο τον ε, την Ευρώπη. Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν πετσοκοπεί λόγω των νέων φιλελεύθερων πολιτικών και πολιτικών λιτότητας που προωθούν όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ μέσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά στην ιστορία του καπιταλισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό παρά την αύξηση των κερδών στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια. Αντί λοιπόν να επενδύεται αυτός ο πλούτος, είτε τον συσσωρεύουν είτε τον παίζουν στις ε, χρηματαγορές. Γι' αυτό ακριβώς η κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτοί να έχουν τον λόγο του εάν θα υπάρξει η επένδυση ή όχι. Αλλά η απάντηση της Κομισιόν είναι να βασιζόμαστε ξανά σε αυτούς τους κερδοσκόπους και μόχλευση μας λένε με ομόλογα έργων. Μα ε, έτσι δεν ε, μοιραζόμαστε το ρίσκο με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας παίρνει τα κέρδη και ο δημόσιος το ρίσκο. Πρέπει να υπάρξουν μαζικές και άμεσες δημόσιες επενδύσεις. Δεν υπάρχει φτώχεια, αν δούμε του συνολικούς πόρους στην Ευρώπη. Οι πλούσιοι έχουν συσσωρεύσει 3-3 εκατομμύρια ευρώ οι μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούμε να πάρουμε αυτό τον πλούτο και να τον επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε δουλειές και υποδομές. Ευχαριστούμε κύριε Μέρφη. Τώρα θα παρέμβουν οι ομιλητές προσωπικά. Καταρχήν θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιβαήλο Κάλφιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ με τη σειρά μου τον εισηγητή. Νομίζω πως κυρία Καρδία Σάβαλ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και τα συμπεράσματά της θα τα δεχτεί η Κομισιόν και ε, τα νομοθετικά σώματα. Έχουμε πει πολλές φορές πως χρειαζόμαστε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα γιατί αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού αλλά δεν θα αντικαταστήσουν τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή ε, λίγο πάνω από το 1% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εμπλέκεται σε χρηματοδοτικά τέτοια μέσα. Έχουμε καλή πρακτική αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να την επανεξετάσουμε και να την αναπτύξουμε στο μέλλον. Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν περιορισμένη χρήση. Κανονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα τα οποία είναι εμπορικά ελκυστικά για να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, αναποτελεσματικότητες αγοράς ε, και για να δημιουργήσουν μόχλευση για τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αλλά και πάλι μιλάμε για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θα ήθελα να αναφέρω τα πολύ καλά παραδείγματα όπου χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα για έρευνα, καινοτομία, μικρομισές επιχειρήσεις και θεωρώ πως πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτά. Πρέπει λοιπόν, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, να έχουμε λιγότερα και πιο εστιασμένα χρηματοδοτικά μέσα και θα ήθελα να πω πως δεν χρειάζεται να τα ρυθμίσουμε υπερβολικά. Πρέπει να αυξηθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια ex post, αλλά δεν μπορούμε να επινοήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά τους εκ των προτέρων, γιατί ε, δεν θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Τέλος, τρία πράγματα τα οποία στηρίζω ε, τυποποιημένες πλατφόρμες όπου μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μαζί με τα ιδιωτικά κονδύλια. Συνεχής επανεξέταση των συμπράξεων αυτών και τέλος ε, η χρήση των ελευθέρων ροών που θα προκύψουν από αυτά πίσω για τον ίδιο σκοπό. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Βόν έχει το λόγο. momento que no diré como dijo anteriormente el comisario. Δεν ξέρω, μάλλον είναι απόν. Εν πάση περιπτώσει, για δύο λεπτά, ο κύριος Κορτές ε, Λάστρα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, αυτό το, για αυτή την έκθεση που στέλνει ένα στεναρό μήνυμα. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα ως προς την αποδοτικότητά μας. Επειδή εργαζόμαστε για τη μελλοντική πολιτική ανάπτυξη, μας ανησυχούν οι περικοπές στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 525 εκατομμύρια θεωρούν ότι η πολιτική αυτή χρειάζεται μέσα καθαρά καινοτόμα, όπως τα μεικτά έσοδα, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και απόδοση. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τα νέα μέσα χρηματοδότησης ώστε να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, διότι διαφορετικά θα θρηνήσουμε θύματα από τη φτώχεια. Και αυτό αφορά και τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα πρέπει να προωθηθεί. Ευχαριστούμε, Ρικάρντο. Τώρα έληξε αυτός ο γύρος και θα λάβουν το λόγο με στα πλαίσια του Catch the Eye, οι ομιλητές που το επιθυμούν. Δίνω το λόγο στην αγαπητή φίλη Ελένα Μπασέσκου. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τέτοια χρηματοδοτικά μέσα. Είναι πολύ ευεργετικό και θα προωθήσει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητά τους έτσι ώστε να φτάσουμε στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης. Πιστεύουμε ότι τα καινοτόμα αυτά μέσα θα διασφαλίσουν μία ε, ευφυή ανταγωνιστικότητα. Όμως η αύξησή τους θα πρέπει να οδηγήσει στην άρση πολλών προκλήσεων από, πλευραν, από πλευράς κυβερνήσεων. Γι' αυτό το νομικό πλαίσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να είναι απλό, απλουστευμένο. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την δελεαστικότητα των χρηματοδοτικών μέσων για τη συνδρομή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Ο κύριος Ζωάου Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το πρώτο μέσο της δεκαετίας του 90 η Επιτροπή διενέργησε έρευνες όπου έγινε λόγος για την συνοχή κυρίως. Μιλούσαμε για προϋπολισμό του 2% του ΑΕΠ. Δεν ξέρω, αλλά αυτές τις μελέτες μπορείς να τις βρείτε ξεχασμένες σε κάποιο σιρτάρι. Μετά από τη μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προϋπολογισμός βρίσκεται στο ίμιση αυτού του ποσού και ε, αποζητάται και η μείωσή του, η περαιτέρω μείωσή τους. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να έχουμε, με ποιο θαύμα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα μέσα. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και οδηγούν σε προβλήματα, γιατί βλέπουμε ότι έχει αποτύχει η πολιτική συνοχή σε κάτι το οποίο αναγνωρίζει και η έκθεση. Τα μέσα αυτά στην ουσία δημιουργούν διχογνωμίες και κρύβουν τους πραγματικούς κινδύνους και μονοπάτια που θα έπρεπε να προωθήσουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Πασκά. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω γνωμοδοτή λέγοντας ότι η παρούσα δομή πορών από τα τρέχοντα χρηματοοικονομικά ε, εργαλεία και προγράμματα είναι δύσκολη, είναι σύνθετη και ασαφής. Πολλοί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν τα όργανα αυτά, αλλά δυσκολεύονται να καταλάβουν τη δομή τους. Θεωρώ ότι ο καλύτερος συντονισμός και ο ε, εξορθολογισμός των εργαλείων αυτών, όπως επίσης και των διαρθρωτικών ταμείων, είναι, ε, είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Τα χρηματοοικονομικά μέσα βρίσκονται βρίσκονται στην υπηρεσία των δραστηριοτήτων των διαφόρων παραγόντων. Γι' αυτό θα πρέπει να, υπάρχει καλή και ενημέρωση και διαφάνεια γύρω από αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια θηρίδα όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ε, έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη στις δραστηριότητές τους. Και τέλος, αν θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι δήμοι να υποφεληθούν από αυτά τα μέσα, θα πρέπει να υπάρξει μια παροχή, μια, να υπάρχουν υπηρεσίες περί αυτών ώστε να γνωρίζουν τον πιο αποτελεσματικό ε, ε, συνδυασμό αυτών των εργαλείων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούχαν έχει τώρα το λόγο, τελευταίος ομιλητή. Ευχαριστώ. Τα χρηματοδοτικά καινοτόμα μέσα έχουν μεγάλη σημασία για να φτάσουμε στους στρατηγικούς στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι όμως ότι δεν έχει οριστεί το πεδίο εφαρμογής αυτών των μέσων. Μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγέ έμπρακτα και περιοριζόμαστε στα, στα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια. Θεωρώ ότι αυτά τα καινοτόμα μέσα θα πρέπει να οδηγήσουν σε ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη συνέργεια των ΜΜΕ και στην ανάπτυξη και έρευνα μέσω συγκεκριμένων μέσων χρηματοδότησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε εκστρατείες πληροφόρησης σε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι έχει το λόγο για να αντιδράσει και να απαντήσει στις ε, παρεμβάσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα σχόλια. Από ό,τι ακούω από τα δικό σας τα σχόλια. Έχουμε μια θετική υποδοχή για την σημασία της, των χρηματοδοτικών αυτών μέσων ε, στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Υπάρχουν ξεκάθαρες ανάγκες και περιορισμοί στον προϋπολογισμό. Οπότε υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από αυτά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία έχουν εν μέρη δοκιμαστεί, αλλά εν μέρη θα δοκιμαστούν και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και υπό ορισμένους όρους και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η όρη στον λεγόμενο αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε δύο πράγματα. Το ένα αφορά την απλοποίηση κατά το οποίο ζητούν όλοι και το δεύτερο είναι ένα τελείως νέο κεφάλαιο και αφορά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Δηλαδή κάποιοι κανόνες για το πώς θα σχεδιάσουμε, θα υιοθετήσουμε, θα εφαρμόσουμε και θα ελέγχουμε την εφαρμογή των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Και μιλάω και για τις δύο αρχές του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο, δηλαδή τα κρατημέλη και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εξαιρετική σας δουλειά πάνω στο περίπλοκο αυτό αντικείμενο. Όπως είπα δεν έχουμε άλλη επιλογή και πρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τον λόγο για δύο λεπτά έχει η κυρία Γκάρδια Θάμπαλ για να τελειώσουμε με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκι. Δεν έχω πολλά να προσθέσω μετά από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των καινοτόμων μέσων για το επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Έγινε λόγος για απλούστευση, για ευφυή μέσα και για εκστρατείες πληροφόρησης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Στην έκθεση λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται ε, επεξήγηση και διαλεύκανση έτσι ώστε και η ΜΜΕ και το τραπεζικό σύστημα να ξέρουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα καινοτόμα μέσα. Επίσης θα ήθελα να διασαφηνίσω ε, κάτι γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα. Υπάρχουν τρία σενάρια ε, επένδυσης, δηλαδή το άριστο όπου υπάρχουν ε, χαμηλή κίνδυνη, χαμηλή επισφάλεια και μπορεί να γίνει άμεση χρηματοδότηση. Μια άλλη κατάσταση όπου αντιμετωπίζουμε ε, ένα project με προστιθέμενη αξία χωρίς όμως να υπάρχει απόλυτη διασάφηση ως προς τους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν μέσω πρόθεσμα, να δούμε ποια είναι η απόδοση, η οποία μερικές φορές δεν είναι επαρκής για να μπορέσουμε να κινηθούμε στις κεφαλαίες Γι' αυτό σε καμία περίπτωση τα μέσα δεν υποκαθιστούν τις επιδοτήσεις ούτε μπορούν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της αγοράς. Θα ήθελα να πω επίσης όπως είπε και ο κύριος ε, Μερφέ, οι ιδιωτικές ε, επενδύσεις έχουν μειωθεί. Δυστυχώς και βλέπουμε ότι στις κεφαλαιογορές υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία. Αυτά τα μέσα όμως αυτό θέλουν να αποδιώξουν έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ε, βιώσιμα σχέδια τα οποία να αποφύγουν την κερδοσκοπία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια Κλείνοντας τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για την πρωτοβουλία σου και ο παππούς σου πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή για να δώσει μεγάλη αγώνα, μεγάλο αγώνα κατά του φασισμού και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι άξια συνεχιστής. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Το επόμενο θέμα είναι η δήλωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Και νομίζω ότι έχει προσέλθει, είναι εδώ ο Επίτροπος Σέπκοβιτς, ο οποίος και θα μιλήσει εξ ονόματος Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, ο Επίτροπος. Now it works. Ξεκίνησα με τη δήλωση ότι η στρατηγική του Δούναβ είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 14 χώρες, 8 ε, κράτη-μέλη και 6 μη κράτη-μέλη με πολλά εκατομμύρια κατοίκους. Από τότε που εισήχθη η στρατηγική έχουμε πιστεί έτσι περαιτέρω για την